Αρχέ μου έστειλαν ένα αίτημα για άρση τη ασυλία του κυρίου Θεοδόρου Ζαγοράκη. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές μου έστειλαν δύο αιτήματα για άρση ασυλία του κυρίου Ούντο Φόκτ. Με βάση το άρθρο 9 του κανονισμού, τα αιτήματα αυτά θα αποσταλούν στην νομική επιτροπή.